Policy Service. I'm for the first the Okay, Thank you. Liebe Kolleginnen Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 9 και 3 λεπτά, οπότε να ξεκινήσουμε. Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω να θέλει κανείς να τροποποιηθεί. Εγκρίνεται λοιπόν. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Πρώτον, η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται ζωντανά στο ίντερνετ, οπότε σας παρακαλώ να μιλάτε με ένα λογικό ρυθμό για να μπορεί να λειτουργεί και η διερμηνία και για να ε, μπορούν να σας καταλαβαίνουν τόσοι ή ε, Και χαιρετίζω όλους τους επισκέπτες μας από το Λισαβόνα, το Λίνεμπουργκ, το Παλέρμο και το Ελσίνκι να υπενθυμίσω ότι το απόγευμα θα έχουμε μία συζήτηση συγγνώμη στις, ε, την Τετάρτη 18, 3 με 6.30 ε, μία συζήτηση με επικεφαλής την κυρία Ζάιφη για τη συνεργασία με τις χώρες του κόλπου που είναι η αντιπρόεδρός μας και η συγκίτρια για τα κράτη του κόλπου. Οπότε να περάσω στο σημείο 3. Η κατάσταση των ε, τριμερών διαλόγων. Κατάσταση πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα έχουμε μία νέα μέθοδο υπολογισμού, που αποφασίστηκε από τον εισηγητή μας ε, στη 3η Οκτωβρίου. Οπότε να του δώσω το λόγο να μα εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Κύριος Τσίκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Αν μου το επιτρέπετε, ήθελα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση μιας ε, ε, σύγκρισης της πρότασης της Κομισιόν του Νοεμβρίου του 2016 που τροποποιεί το άρθρο 2.7 του, κανονισμού, του βασικού κανονισμού καταπολέμησης του ντάμπινγκ ε, στο κομμάτι όπου αναφέρεται στη διάκριση μεταξύ χωρών με οικονομία αγοράς και χωρών χωρίς οικονομία αγοράς όπου η κανονική ε, τιμή ε, καθορίζεται βάση μιας χώρας αναφοράς. Ε, το πρωτόκολλο προσχώρηση της Κίνας στον ΠΟΕ το 2001 άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ε, περιοριστικής ερμηνείας. Η μη συμμορφώση λοιπόν ε, του σημερινού κανονισμού στο άρθρο 2.7 με τις αρχές και τους κανόνες του ΠΟΕ ισχύει. Η νέα πρόταση υπερβαίνει αυτή τη διάκριση αφήνει μια διάκριση μεταξύ χωρών ΠΟΕ και χωρών που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ. Έτσι επιλέγεται η εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας. Η πρόταση εισάγει στο νέο άρθρο 2.6 τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιηθεί η τυπική μεθοδολογία για τις χώρες του ΠΟΕ, αλλά μια νέα μεθοδολογία εναλλακτική. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και εφόσον παρατηρηθούν σημαντικές τρευλώσεις στην τρίτη χώρα. Να υπενθυμίσουμε λίγο την αρχική αξιολόγηση εκ μέρους της ε, Επιτροπής μας, εκ μέρους όλων των ε, συναδέλφων. Αρχικά υπήρξε κάποια σύγχυση, κάποια καχυποψία, μια δυσπιστία και διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τα βασικά στοιχεία της πρότασης. Καταφέραμε, πιστεύω, μέσω της συνεργασίας να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα, να κάνουμε καλή δουλειά με διάφορες προτάσεις, ε, συμμετοχή, εκτίμηση, δυνατότητα διαμεσολάβησης, ε, ώστε να καταλήξουμε σε μια συνένεση αρκετά ευρεία ώστε να δεχθούμε την πρόταση αυτή ολοκλήρωσης επικεντρωμένη πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία. Από την Κομισιόν μέχρι το Συμβούλιο, μέχρι την Επιτροπή ΙΝΤΑ, όλοι οι συνάδελφοι ε, χρησιμοποίησαμε μία νέα προτεραιότητα, το να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το πιο αποτελεσματικό δυνατό μέτρο για την προστασία της βιομηχανίας στην Ευρώπη ενώπιον της, ε, του αθέμητου ανταγωνισμού. Οι εργασίες ε, του Κοινοβουλίου και να υπενθυμίσω το πλαίσιο στο Συμβούλιο όλα πήγαιναν καλά, ε, συμφωνούσαν με ό,τι πρότεινε η Κομισιόν. Εμείς στο Κοινοβούλιο εμπλουτίσαμε τη λίστα των κριτηρίων που καθορίζουν ε, τη σημαντική στρέβλωση της αγοράς ως ορισμό. Αναφερθήκαμε στο ε, τραπεζικό δίκαιο, στο δίκαιο ε, ε, της χρεοκοπίας και μιλήσαμε και για την μισθολογική ισότητα. Και να κάνω εδώ μια παρέθεση, για πρώτη φορά συμπεριλάβαμε την κοινωνική πτυχή. Πιστεύω ότι δώσαμε δομή και ισχύ στην έκθεση της Κομισιόν για τις τρίτες χώρες που αποτελεί θεμελιώδη στοιχείο ολόκληρου του οικοδομήματος και περιλαμβάνει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζεται η βιομηχανία. Μην ξεχνάμε ότι η έκθεση της Κομισιόν περιλάμβανε διακριτική ευχέρεια ως, τη διακριτική ευχέρεια ως έννοια δεν ήταν υποχρεωτική εμείς συμβάλαμε ώστε ε, να γίνει υποχρεωτική δηλαδή τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σήμερα αποτελούν ε, συγκεκριμένη απτή απόδειξη και εμείς ε, προσθέσαμε ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί οτιδήποτε επιπλέον ως βάρος για τη δική μας βιομηχανία ε, και κυρίως όσον αφορά το βάρος της απόδειξης. Διότι από το κείμενο έτσι όπως έχει με τη συγκεκριμένη θεολογική σκέψη ε, δώσαμε να καταλάβουν όλοι ότι ε, το να αποδείξει κανείς ότι ορισμένα κόστη δεν αποτελούν στρέβλωση δεν θα βαραίνει τις δικές μας επιχειρήσεις. Ε, Συμμετείχαμε κάποιου μηχανισμού, ε, δημιουργήσαμε κάποιου μηχανισμού στο κείμενο και στη διακήρυξη τη Κομισιόν που ε, επισυνάπτεται στο κείμενο παρέχεται η δυνατότητα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να διατυπώσουν μια θέση, μια αξιολόγηση, να συμβάλλουν όσον αφορά καταστάσεις που έχουν τελματώσει, ε, όπου δεν υπάρχει έγκαιρη επαλήθευση και επακριβής ε, δηλαδή ένας συγκεκριμένος ρόλος του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που μπορούν να παρέμβουν φυσικά μέσω του διαλόγου, μέσω μιας συνομιλίας που εφόσον ε, χρειαστεί θα ανταποκρίνεται καλύτερα όσον αφορά την εξέβεση της πιο αποτελεσματικής μεθόδου. Ε, στα ε, αιτιολογικές σκέψεις θέλουμε ορισμένα κομμάτια να συμπεριληφθούν, να μεταφερθούν στο βασικό κείμενο ώστε να υπάρχει μια πλήρης και αποτελεσματική ε, εκτίμηση της κατάστασης με ε, την ίδια οργάνωση όσον αφορά όλες τις περιπτώσεις μέσα στο κείμενο. Τι επιτύχαμε. Για πρώτη φορά, και αυτό θεωρώ είναι εξαιρετικό, για πρώτη φορά στην εμπορική νομοθεσία συμπεριλαμβάνονται ε, κοινωνικο-περιβαλλοντικά στοιχεία, τα οποία από τη μια πλευρά έχουν πολιτική αξία, από την άλλη όμως ε, προσδίδουν και σημαντική αποτελεσματικότητα στον καθορισμό της κανονικής αξίας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η αλλαγή υπήρξε πολύ σημαντική. Τέλος, ε, καταφέραμε να βρούμε μία διατύπωση για το βάρος της απόδειξης που απέτυχε, θυμίζω, έναν τριμερή διάλογο επιπλέον, ο οποίος ωστόσο κατά την κρίση μου μας βοήθησε να πραγματοποιήσουμε ένα βήμα μπροστά, μια αλλαγή που μας αφήνει πιο ικανοποιημένους ε, σε σχέση με την έκβαση των εργασιών μας. Συνοπτικά λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ε, ένα κείμενο πιο σαφές, ε, πιο αξιόπιστο, το οποίο στην τελική του μορφή έλαβε και την υποστήριξη ολόκληρης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που ε, βοηθά στην εφαρμογή του εργαλείου αντι-dumping ε, και βιομηχανία η οποία έπαιξε πολύ επικριτική για την αρχική πρόθεση της Κομισιόν. Χάρη στους μηχανισμούς που έχουν συμπεριληφθεί θα μεριμνήσουμε για μια ε, αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας αντι-dumping από το 2018. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη σοβαρότητα για την αφοσίωσή σας, ε, για την επικοδομητική συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς και ευχαριστώ ιδιαίτερα εσάς κύριε ε, Πρόεδρε, κύριε Λάγκα, για το εξαιρετικό σας έργο ε, καθώς εσείς υπήρξατε, πώς να το πω, ο διαχειριστής όλου αυτού του εκπληκτικού αποτελέσματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να σας απευθύνω με τη σειρά μου τις δικές μου ευχαριστίες. Ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό με την αναγκαία αφοσίωση και επιτύχαμε καλά αποτελέσματα. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ. Συνολικά λοιπόν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να είναι περήφανο για αυτά που επιτύχαμε για αυτό το νομοθέτημα. Λοιπόν, τα κείμενα υπάρχουν, ήδη έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας. Θα ψηφίσουμε το κείμενο και όπως είπε ο εισηγητής υπάρχουν κάποιες ε, συμπληρωματικές διευκρινήσεις και μια επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι επίσης δημοσιευμένα τα κείμενα αυτά. Υπήρχε και ένας δεύτερος τριμερής διάλογος ο οποίος αυτή τη στιγμή βέβαια ίσως να μην ε, διεξάγεται αλλά υπάρχει. Είναι ο τριμερής διάλογος για τον εξυγχρονισμό των μέσων ε, εμπορικής προστασίας αλλά μέχρι στιγμής ε, δεν διεξάγεται με πολύ ζωηρότητα. Η Εσθονική Προεδρία θα κάνει μια νέα προσπάθεια στις 18 Οκτωβρίου θα υπάρξει ένας ε, ε, επιπλέον τριμερής διάλογος για αυτό το θέμα έτσι τουλάχιστον δήλωσε η Εστονική Προεδρία και δήλωσε ότι έχει κάθε βούληση να κλείσει το θέμα μέχρι τέλος του έτους. Να δούμε αν θα το επιτύχει. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσω λοιπόν στο σημείο 4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπάρξει μια ε, παγκόσμια συμμαχία για το εμπόριο ε, μέσων βασανιστήριων. Η διαδικασία ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη και βασίζεται και στα νομοθετήματα που έχουμε εγκρίνει τα τελευταία χρόνια. Η συγγήτριά μας ήταν η Μαρίτ Σιάκη. Να της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί έχω την ευκαιρία να δω, να δούμε όλοι πόσο η δουλειά μας αναβαθμίζει την ε, νομοθεσία κατά των βασανιστήριων. Και αυτό έχει οδηγήσει και σε πολυμερείς πρωτοβουλίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπλέκοντας την Αργεντινή και τη Μογγολία μεταξύ άλλων. Στην εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Επίτροπος Μάλστρομ είχε την ευκαιρία μαζί με εμπειρογνώμονες αλλά και θύματα ε, βασανιστήριων να ξεκινήσει αυτή τη συμμαχία για το ελεύθερο εμπόριο χωρίς βασανιστήρια, μια συμμαχία την οποία θέλουμε να διπλωμάτες και υπουργοί από 59 ε, χώρες που έχουν, που έχουν υπογράψει ε, τα καταστατικά έγγραφα αυτής της συμμαχίας. Ήταν μια πολύ ισχυρή εκδήλωση που έδειξε πόσο εμείς θέλουμε να ανεβάσουμε το πύχη και πόσο θέλουμε να υιοθετήσουμε εμπορικούς κανόνες που που παρεμποδίζουν τα βασανιστήρια και αυτό θα έχει πραγματική αλλαγή στη ε, ζωή των ανθρώπων. Ένας μίλησε για τον πατέρα του που βασανίστηκε μέχρι ε, θανάτου πριν γεννηθεί ο ίδιος, ενώ μια άλλη ε, γυναίκα μίλησε για τα βασανιστήρια που είχε υποστεί ως παιδί στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ε, αυτές οι εκδηλώσεις απλά αποτέλεσαν εκδηλώσεις έναρξης αυτής της εκστρατείας για τη συμμαχία και ελπίζουμε εμείς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνουμε τη διαφορά, να μεγαλώσει η συμμαχία, να πείσουμε όλες τις χώρες να υπογράψουν για αυτή τη συμμαχία για ένα εμπόριο ελεύθερο βασανιστήριων και ενδεχομένως να ξεκινήσουμε να ε, σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο σε λίγα χρόνια να υιοθετηθεί μια πρωτοβουλία από σύσσωμο των ΟΗΕ, για παράδειγμα μια ε, διεθνή συνθήκη ή σύμβαση για το θέμα αυτό. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορώ να σας πω και περισσότερο, το βασικό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε ηγετικό πνεύμα και προσπάθησε με επιτυχία να μεταφέρει τα πρότυπά μας ε, σε μια διεθνή πλατφόρμα που να εμπλέκει και άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Η Χίλντε Χάρντεμαν. Έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Συμφωνούμε, κυρία Χάκα, με την αξιολόγησή σας η έναρξη της ε, συμμαχίας αυτής, η κήρυξη της έναρξης ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε πραγματικά το πνεύμα ηγεσία που τη διέπει. Είχαμε εκπροσώπους από τα 58 κράτη που συμφώνησαν να προσχωρήσουν στην Παγκόσμια Συμμαχία, εκπροσώπους από διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πράγματι ανθρώπους που έχουν νιώσει στο πετσί τους ε, το, ε, τα βασανιστήρια αυτά και ε, αποτέλεσαν και εξέφρασαν τις μαρτυρίες άλλων που έχουν πληρώσει με την ίδια τους τη ζωή ε, τα βασανιστήρια. Ε, όπως είπε και η Επίτροπος Μάλστρομ, ε, παρέστησαν εκπρόσωποι από διάφορα κράτη για να στηρίξουν τη συμμαχία και να τονίσουν πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε ο ένας πλάι στον άλλον σε αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, εσάς προσωπικά, αλλά και την Επιτροπή Ίντα για την στήριξη που μας δώσατε στη Νέα Υόρκη σε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στη στήριξή σας για να καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες και να παρακινήσουμε και τρίτες χώρες να υιοθετήσουν παρεμφερή νομοθεσία. Οι παρούσες χώρες ανέλαβαν την ευθύνη να συντάξουν δικιά τους ε, νομοθεσία για τον περιορισμό ενδεχομένως στην απαγόρευση των ε, αγαθών, των προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως σε βασανιστήρια. Να συντάξουν σε κάθε περίπτωση νομοθεσία κατά των βασανιστήριων και το σημαντικό είναι πώς τα υφιστάμενα εξωτερικά προγράμματα μπορούν να αξιοποιηθούν στην εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού για το εμπόριο ελεύθερο βασανιστήριων και να στηρίξουμε τις χώρες που θα αναλάβουν αυτή τη δέσμευση και εμπορικά. Θέλουμε ε, πολιτική στήριξη για να διευρυνθεί η συμμαχία και αυτή η πολιτική στήριξη είναι αδύρυτη ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, στόχος μας είναι ο εξής. Θέλουμε να διευκολύνουμε την παροχή τεχνικής βοήθειας, την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών μελών της Συμμαχίας και προσπαθούμε να προβλέψουμε τη διοργάνωση ενός εργαστηρίου όπου θα υπάρχουν και θα παραστούν εμπειρογνώμονες από τα διάφορα κράτη-μέλη στις Βρυξέλλες το πρώτο εξάμεινο του 2018 και θέλουμε και στοχευμένη τεχνική βοήθεια να μπορέσουμε να δώσουμε. Η πολιτική σας στήριξη είναι εξαιρετικά πολύτιμη, είναι ανεκτήμητη. Θα σας τηρούμε ενήμερους για τα επόμενα βήματα τα δικά μας και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Βεβαίω θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τι εργασίε σα και ελπίζουμε να σα βοηθήσουμε. Όπω πρότεινε η Μαρίτια Σχάκε για να είναι πραγματικά πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Και χαίρομαι που και για άλλο ένα θέμα η Ένωση παίζει τον πρωτοπόρο ρόλο, θέτει το θέμα εμπορίου που να βασίζεται σε αξίες. Ορισμένοι επικρίνουν διαρκώς την εμπορική πολιτική της Ένωσης, αλλά πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι με βάση τα νομοθετήματα και την πολιτική μας και με βάση κυρίως ε, τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ξεκινήσει μια πολιτική στον τομέα του εμπορίου που να βασίζεται σε αξίες. Και αυτό είναι ένα εξαίρετο παράδειγμα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί μέσω της εμπορικής πολιτικής να βοηθήσει ουσιαστικά τους πολίτες. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και την κυρία Χάλντεμα. Να περάσουμε στο σημείο 5. Στις 13 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε στην εμπορική πολιτική και την ε, αποκάλεσε πρώτη προτεραιότητα στην ομιλία του κυρίου Γιούγκερ για την κατάσταση της Ένωσης και ανήγγειλε μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες θα συζητήσουμε ε, σε διάφορες συνεδριάσεις. Και μεταξύ αυτών των ε, πρωτοβουλειών είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων ε, της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου. Υπήρχε ήδη αυτό και με μια ανακοίνωση ε, που υπήρξε στην αρχή του χρόνου έχουν γίνει πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Δηλαδή, πώς έχουν τα πράγματα. Από τη μία η παγκοσμιοποίηση μας φέρνει αντιμέτωπους με ε, προκλήσεις. Υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Είχαμε χαιρετήσει αυτή την ανακοίνωση και τώρα περιμένουμε για να δούμε πώς θα συγκεκριμενοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε εδώ τον Ιώζεπ Κόρτε, τον παλιό μας γνώριμο, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σα μιλήσω σύντομα σήμερα το πρωί για το ενεμπορική δεσμη μέτρων, ε, όπω αναφέρθηκε στην κατάσταση τη Ένωση. Έχει πέρασει ένα μήνα σχεδόν από την ομιλία εκείνη του Πρόεδρου Γιούνκερ και πράγματι το εμπόριο υπήρξε σημαντικό κομμάτι τη ομιλία, η οποία όχι μόνο υπήρξε εξαιρετική, αλλά υπήρχε και κάτι ενδιαφέρον ότι η Κομισιόν ταυτόχρονα την ίδια μέρα πρότεινε μία δέσμη μέτρων, μία δέσμη προτάσεων. Οκτώ προτάσεις ήταν αυτές. Θα σα τι παρουσιάσω εν συντομία λίγο αργότερα. Όπως είπατε εσείς κύριε Λάγκε, αποτελούν τις ε, τελευταίες ε, απόψει της Κομισιόν για την παγκοσμιοποίηση και αποτελούν και τη δική μα απάντηση για τόσα συμβαίνουν γύρω μας στον κόσμο. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα, όπου εμφανίζονται νέες προκλήσεις. Δίνει και μια απάντηση ε, για τα όσα έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια όπου η εμπορική πολιτική είχε αποτελέσει ένα επίμαχο θέμα και όλο αυτό αποτελεί και ένα follow-up στο εγγραφό προβληματισμού που παρουσίασε το Μάιο ή για την παγκοσμιοποίηση κομισιών γενικότερα. Είναι λοιπόν μια σημαντική δέσμη μέτρων, μια καλή ομιλία και όλες αυτές αυτή τη στιγμή περνούν από το σύστημα φυσικά και από το κοινοβούλιο. Σήμερα σκοπός είναι μάλλον να καταδείξουμε την βασική, τη θεμελιώδη φιλοσοφία. Οκτώ λοιπόν μέτρα προτάθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου, τρεις ε, συστάσεις για διαπραγματευτικές ε, ε, οδηγίες, σχέδια εντολών όπως αναφέρθηκαν, για την Αυστραλία, για την Νέα Ζηλανδία και για το Πολυμερές Δικαστήριο Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών. Υπήρξε και μια ανακοίνωση ε, που βασίζεται σε μια πολιτική ε, σκέψη και υπάρχει μια σημαντική έκθεση προόδου για το ε, εμπόριο που παρουσίασε η κυρία Μάλμστρομ πριν από δύο χρόνια και υποσχέθηκε απολογισμό μετά από δύο χρόνια κάτι που έχει συμβεί. Πρέπει να πω ότι αυτό το έγγραφο παραμένει βασικό έγγραφο πολιτικής του Επιτρόπου μου για της Επιτρόπου μου για την εμπορική πολιτική και υπάρχει και μια σημαντική νέα πρόταση για την ε, σύσταση μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα πρέπει να προσφέρει αρρωγή στην Κομισιόν για τι διαπραγματεύσει στον τομέα τη εμπορική πολιτική. Και τέλο, υπάρχει μια γενική ανακοίνωση που ονομάζεται ισορροπημένη και ολοκληρωμένη εμπορική πολιτική για την Τιθάσευση της παγκοσμιοποίηση Το έγγραφο αυτό ουσιαστικά αποτελεί το ραχοκοκαλιά της πολιτικής. Ε, αναφέρει τα επτά ε, βασικά σημεία μαζί σε ένα συνεκτικό κείμενο εκφράζοντας μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Πολλά λοιπόν ε, πράγματα έχουμε μπροστά μας όσον αφορά νέες ιδέες, νέες προτάσεις και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ε, σημερινή ατζέντα που ήδη υπάρχει και ήδη τρέχει τις διαπραγματεύσεις για τις διάφορες συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών με τις χώρες Μερκοσούρ, με το Μεξικό, που δεν ε, προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν πολιτικά μέχρι τα τέλη του έτους. Έχουμε την ε, συμφωνία με την Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, την Ιαπωνία. Είναι μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα. Δεύτερον τώρα ας προσπαθήσω, αν μου επιτρέπετε, να σας ε, ξεναγήσω λίγο στις ε, ε, πολιτικές απόψεις στις οποίες βασίζεται η δέσμευτη προτάσεων. Η Επιτροπή φυσικά αναγνωρίζει ότι το εμπόριο δεν είναι αυτός σκοπός είναι μια βασική κινητήριο δύναμη για μια ανταγωνιστική ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που ευημερεί. Θα έχετε ξανακούσει πάνω από 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας υποστηρίζονται από τις εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο. Μια παγκοσμιοποιημένη λοιπόν οικονομία δεν πάβει να αποτελεί κάτι αποφελές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους καταναλωτές και τους πολίτες της. Εκεί εμφανίζονται κάποιες ε, νέες ιδέες μέσω αυτής της νέας δέσμης. Το νέο εμπόριο πρέπει να έχει διαμορφωθεί ε, προορατικά και θα πρέπει να το μοιραζόνται όλοι. Θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιες αξίες και σε κάποιο σύστημα κανόνων. Ο ίδιος ο πρόεδρος πολύ συχνά χρησιμοποίησε ε, την έκφραση «η Ευρώπη που προστατεύει». Η Ευρώπη δεν είναι αγαθή. Είμαστε ανοιχτοί, είμαστε ανοιχτόμυαλοι, αλλά δεν είμαστε αγαθοί. Για όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει ένα ανοιχτό εμπορικό σύστημα βασισμένο σε κανόνες με τον ΠΟΕ στο επίκεντρό του. Και σε περίπτωση προστατευτισμού η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να ηγηθεί. Αυτό, έγινε χθες, αυτό είναι που έκανε χθε η κυρία Μάλνστρομ προετοιμάζοντα ε, την διάσκεψη του Μπονοσάιρε, του, ε, MC11 για τα τέλη του έτου. Ο πρόεδρος Τραμπ, ε, ο πρόεδρος Μπούς είπε, κατάλαβε ο κύριος ε, ομιλητής, ο κύριος Τραμπ δεν ανέφερε ούτε μία φορά το Brexit. Είναι σαφές ε, ότι οι προκλήσεις αυτές αποτελούν, χαρακτηρίζουν οποιαδήποτε ενέργειά μας. Όπως είπα προηγουμένως, ε, οι προτάσεις ε, σε τελική ανάλυση καταλήγουν ε, στο έγγραφο Trade for All της Σισίλια Μάλμστρομ, εμπόριο για όλους, που ε, δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2015. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για να λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίε εξελίξει και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Αλλά οι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Εμπορική Στρατηγική παραμένουν οι ίδιε. Αγωνιζόμαστε για ανοιχτό εμπόριο βασισμένο σε κανόνε που να υποστηρίζει την ευημερία μα, που να υποστηρίζει τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά, καταναλωτικά, κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, καθώ και στον τομέα τη προστασία τη εργασία και ε, για την προστασία των βασικών αξιών τη Ευρώπη. Η έκθεση ε, της 14 Σεπτεμβρίου κοιτά τι έχει επιτευχθεί, τι δεν έχει πάει πολύ καλά ε, εξετάζει τους εμπορικούς προσανατολισμούς που είχαν διαμορφωθεί το 2015 και κοιτάζει και προς το μέλλον. Όσον αφορά το μέλλον, θέλω να επιστήσω την προσέξη σε μια άλλη έκθεση που πρόκειται να κυκλοφορήσει από την Κομισιόν τον Νοέμβριο. Πρόκειται για μια έκθεση ειδικά αφιερωμένη στην ε, εφαρμογή όλων των συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών, των FTA που έχουν συναυθεί μέχρι σήμερα. Η έκθεση αυτή νομίζω τώρα ε, βρίσκεται σε διαδικασία ε, έγκρισης από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα τη δούμε τον Νοέμβριο. Εκεί γίνεται μια αναφορά για κάθε FTA βάσει συγκεκριμένων δικτών και κριτηρίων ώστε να αντιληφθούμε ότι παρότι είμαστε φιλόδοξοι στη διαπραγμάτευση νέων FTA, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτέ που έχουμε ήδη λειτουργούν αυτέ οι συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών και ότι αν δεν λειτουργούν πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Οπότε είναι πολύ καλό που θα εμφανιστεί αυτή η έκθεση, η οποία μάλιστα θα εκπονείται ετησίω. Θέλουμε να έχουμε ετήσιε εκθέσει για την υλοποίηση των συμφωνίων ελευθερών συναλλαγών και αυτέ αποτελούν μια καλή ευκαιρία ώστε το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα και ενδιαφερόμενοι να ε, να παρακολουθούν και αυτοί ε, την υλοποίηση αυτή των συμφωνιών αυτών. Ε, τέλος, θα ήθελα να αναφέρω δύο άλλα σημαντικά ζητήματα. Οι δομές, η αρχιτεκτονική των εμπορικών συμφωνιών πρώτον και δεύτερον η διαφάνεια. Και τα δύο περιλαμβάνονται σε αυτή τη δέσμη. Σε αυτή την επιτροπή πριν από μερικούς μήνες συζητήσαμε ε, τα συμπεράσματα πρέπει να εξάγουμε από την γνωμοδότηση του δικαστηρίου ε, του Μαΐου για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης. Όπως ξέρετε, η απόφαση αυτή επικύρωσε ότι σχεδόν τα πάντα στην FTA της Σιγκαπούρης ε, μπορούν να θεωρηθούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δύο εξαιρέσεις μόνο. ε, ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και την ε, επίλυση διαφορών, επενδυτικών διαφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών. Προσπαθήσαμε να δοθεί επαρκής χρόνος σε εσά και στα κράτη-μέλη να δείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στον καλύτερο δυνατό βαθμό αυτή τη γνωμοδότηση και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την κατάσταση αυτή ώστε να αποφύγουμε προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν όπως τις δυσκολίες με την επικύρωση της ΕΤΑ και πώς να αποκομίσουμε κάποια διδάγματα. Αντιλαμβανόμενοι φυσικά ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα όπου οι υπουργοί και ε, κοινοβούλια ε, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίζουν ε, τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Τι έχουμε κάνει λοιπόν εδώ και με τα κράτη-μέλη, έχουμε παρουσιάσει τι ιδέε μα για μια καλύτερη αρχιτεκτονική μελλοντικών συμφωνίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάσαμε ειδικότερα τι θα κάνουμε με την προστασία των επενδυτών και πού θα τη συμπεριλάβουμε. Πρέπει να πω ότι η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεχίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτό εξηγεί και γιατί αν δείτε την εντολή που έχουμε προτείνει για την FTA με την Αυστραλία και την ε, Νέα Ζηλανδία, εκεί το κομμάτι της προστασίας των επενδυτών δεν έχει συμπεριληφθεί. Αυτό Θέλω να είμαι σαφή. Δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να συμπεριληφθεί στο μέλλον. Απλά προχωράμε ψηλαφιστά με τα κράτη-μέλη, ψάχνοντας να δούμε ε, κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον για να ε, συμπεριληφθεί και αυτό η προστασία ε, των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και των επενδυτών ε, με χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία και αν καταλήξουμε στο αντίστοιχο συμπέρασμα τότε θα υπάρξει ένα δεύτερο σύνολο εντολών από την Κομισιόν που θα καλύπτει τα σημεία αυτά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μας να γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα ε, να δεχθούν να καλυφθούν και αυτοί οι τομείς πολιτικής. Γιατί, διότι αυτά τα κομμάτια των μελλοντικών ε, εμπορικών συμφωνιών θα, θα είναι δύο μορφών. Ή θα έχουμε κλασικές FTA, ε, κλασικές αλλά ε, ε, με ευρύ αντικείμενο, με ευρύ πεδίο εφαρμογής και ανοιχτές, περιλαμβάνοντας και όλα τα στοιχεία προστασία και μετά θα υπάρχει ένα δεύτερο τύπο συμφωνία που θα είναι μια μεικτή συμφωνία η οποία θα καλύπτει και ε, τις ε, ε, επενδύσεις χαρτοφυλακίου και την προστασία των επενδύσεων. Οπότε με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όπως καταλαβαίνετε, να ε, δω και ποια είναι η άποψη εδώ του Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα με την Αυστραλία και την Αζηλανδία. Δεν θέλουμε να περιμένουμε ε, να... Και γι' αυτό έχουμε υποβάλει και τα σχέδια εντολών πίσω από όλα αυτά από πολιτική άποψη και γι' αυτό ε, προχωρά πολύ ε, προσεκτικά σε αυτό το ρευστό τομέα η Κομισιόν είναι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και φυσικά η Κομισιόν ε, δεν θέλει να θεωρηθεί ότι σφετηρίζεται τις εξουσίες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ταυτόχρονα όμως είναι καθήκον μας να δείξουμε ότι η επικύρωση από τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν μπορεί να είναι το, ε, η απότερη δοκιμασία της δημοκρατίας. Η δημοκρατική απόφαση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται από τη συνθήκη πρώτον από εσάς, αλλά και από το γεγονός ότι οι Υπουργοί όταν έρχονται στις Βρυξέλλες ε, είναι απολύτω υπόλογοι. Έχουν λάβει εντολή από τα εθνικά του κοινοβούλια. Αυτό θεωρείται δηλαδή τουλάχιστον. Εκεί δυστυχώ ε, ε, ξεφεύγει λίγο η συζήτηση όταν μιλάμε για το TTIP και τη ΣΕΤΑ και ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι η επικύρωση των κοινοβουλίων είναι η απόλυτη ε, δημοκρατική εγγύηση. Εμείς διαφωνούμε με αυτό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε ε, στις εθνικές κυβερνήσεις τα εργαλεία να τα συζητήσουν αυτά με τα εθνικά κοινοβούλια. Γι' αυτό η διαφάνεια είναι τόσο σημαντική. Και γι' αυτό θέλω να κλείσω για τη διαφάνεια, με τη διαφάνεια ακριβώς η δημοσίευση λοιπόν των σχεδίων εντολής ε, για τις FTA με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία ε, ε, είναι γεγονός και τα έχουμε στείλει αυτά τα σχέδια ταυτόχρονα και στα Εθνικά Κοινοβούλια όπως τα στείλαμε και σε εσά. Όλα τα κράτη-μέλη δεν τα έλαβαν με ιδιαίτερη χαρά. Ωστόσο, η Κομισιόν αισθάνθηκε ότι αυτό ήταν απολύτω απαραίτητο για να δείξουμε αφενό ότι είμαστε απολύτω διαφανεί, ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Και δεύτερον, διότι πολλέ από αυτέ τι ε, εντολέ θα πρέπει ούτω ή άλλω να ληφθούν υπόψη. Και τρίτον, για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη σε όσο το δυνατόν νωρίτερο στάδιο να ξεκινήσουν συζητήσει στα κοινοβούλια του ε, για προτάσει αυτέ τέτοιου είδου από την Κομισιόν. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη ώστε να ε, διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν πλέον συζητήσεις από αρκετά πρώιμο ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια ε, όσον αφορά τις προτάσεις αυτές της Κομισιόν. Αυτό πιστεύω ήταν σημαντικό. Κάτι τελευταίο για τη διαφάνεια. Η δέσμη αυτή προτάσεων συνιστά και δημιουργεί και μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ε, και του τομέα ε, θα ασχοληθεί με τις διαπραγματεύσεις με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και τις διαπραγματεύσεις για τις FTA θα βασιστεί σε διάφορους κανόνες κομισιών στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας του Better Regulation. Αυτό σημαίνει ότι έχει κυκλοφορήσει μια ε, πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να το ετηθούν μέχρι την 1η Οκτωβρίου τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα υπάρξει μια εσωτερική αξιολόγηση εντό τη Κομισιόν για να επιλεχθούν οι καλύτεροι δυνατοί υποψήφοι και ελπίζουμε ότι αυτή η ομάδα θα ξεκινήσει τι εργασίε τη ε, στι αρχέ του 2018. Η ομάδα αυτή δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ε, τον υπάρχοντα διάλογο ε, της κοινωνίας των πολιτών ε, που είχε συναντηθεί την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για μια επιπλέον ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πήρα λίγο παράπονο από το χρόνο σας από ό,τι είχε προβλεφθεί, αλλά πιστεύω ότι παρουσίασα τα βασικά πολιτικά ε, σημεία της δέσμης και ευχαριστώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Um, ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να κάνει ερωτήσεις ή παρεμβάσεις. Α, σχεδόν όλοι. as well. Yeah. And Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα το κατάλογο μιλητών. Θα σας παρακαλούσα όχι πάνω από τρία λεπτά η Ίνμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Κόρτε για τη θαυμάσια συνόψιση της πολιτικής της Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Θέλω να συγχαρώ για τα εξή δύο. Πρώτον, γιατί τέθηκε ως προτεραιότητα η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή η αντιμετώπιση της μέσω της εμπορικής πολιτικής για να επιτύχουμε τους στόχους μας, δηλαδή πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε την ε, παγκοσμιοποίηση. Πρώτο λοιπόν να το αναγνωρίσουμε αυτό ως θέμα. Και δεύτερο ότι αυτό πρέπει να συνοδεύεται με μια αξιολόγηση, όπως έχουμε ζητήσει ως Επιτροπή. Και εγώ προσωπικά έχω επιμείνει να υπάρξει μια σφαιρική αξιολόγηση για το πώς λειτουργούν οι συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου και μάλιστα να ε, εκδίδονται τέτοιες εκθέσεις κάθε χρόνο. Να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα. Πώς θα επιτύχουμε η παγκοσμιοποίηση να μην εξαιρεί κανένα. Δηλαδή να υπάρξει αυτό που αποκαλούμε βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει γίνει καλή δουλειά για το θέμα αυτό, αλλά δεν περιλαμβάνεται καμία δυνατότητα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας μηχανισμός που να βασίζεται σε κυρώσεις. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο. Μας είπατε ότι ε, δεν είχαμε καταλήξει στον ε, μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών επενδυτών κρατών και για, χρειάστηκε γι' αυτό να ξανανοίξει μια κλεισμένη συμφωνία. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι πολίτες. Πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε η ηγεσία στο θέμα αυτό. Πρέπει να υπάρξει ο βέλτιστος μηχανισμός που να βασίζεται σε κυρώσεις. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να μας βοηθήσει και πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου, να ακούγεται η φωνή μας, η φωνή δηλαδή των πολιτών που εκπροσωπούμε και ε, να λαμβάνεται και υπόψη η φωνή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, σε αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων θα υπάρξουν και ειδικοί για τα θέματα ισότητας φύλου, γιατί εάν θέλουμε να μην αποκλείει κανένα η παγκοσμιοποίηση, πρέπει να μην αποκλείονται οι γυναίκες. Χρειάζονται ειδικοί, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την συμπερίληψη ε, με πλήρη τρόπο της προπτικής φύλου. Όλα αυτά είναι βέβαιως καινούργια μέτρα. Προχωράμε για να διαμορφώσουμε το μέλλον. Αλλά τι γίνεται με τις ήδη υπογραφείς σε συμφωνίες που δεν περιλαμβάνουν κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης. Θα μελετήσετε πώς μπορούμε να έχουμε πιο ευέλικτους μηχανισμούς ενημέρωσης αυτών των συμφωνιών για να συμπεριλάβουν ε, κεφάλαια βιώσιμη ανάπτυξη. Γιώχιμ Σούστα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα η εμπορική πολιτική δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένη. Είναι τμήμα της διαμόρφωση των παγκοσμίων οικονομικών σχέσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει καταλάβει. Έχουμε πολύ διαφορετικές συμφωνίες που πολλές φορές ε, αφορούν και άλλους τομείς πολιτικής. Για παράδειγμα, έχουμε τη συμφωνία με την Αφρική, την συμφωνία σύνδεση με την Ουκρανία, όπου η εμπορική πολιτική είναι ένα μόνο τμήμα της επίτευξης γενικότερων στόχων. Αυτό είναι σκόπιμο βέβαια. Αλλά πώς θα προχωρήσουμε, ούτω ώστε να υπάρχει συνέπεια στην πολιτική μα, Ποια θα είναι η βάση της πολιτικής μας. πώς ε, συνδυάζεται η εμπορική πολιτική με την πολιτική συνεργασία μας για την Αφρική. Τι δομές θέλει να δημιουργήσει η Κομισιόν, ούτω ώστε να διασφαλίσει ότι τα καθήκοντα που έχουμε, για παράδειγμα, για μακροοικονομική στήριξη και πληρωμών προς την Ουκρανία, είναι όντως ε, συμβατά με τους εμπορικούς μας στόχους. Θα ήθελα περισσότερη πληροφόρηση γι' αυτό. Δεύτερο, Είπατε ότι θέλουμε να βασίζεται σε αξίες ε, ο μηχανισμός, ε, ο δικαστικός μηχανισμός επίλυσης των διαφορών. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά το θέμα δεν είναι η προστασία των επενδύσεων. Στόχος μας είναι να μην έχουν ειδικά δικαιώματα μόνο οι επενδυτές. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να έχουν και υποχρεώσεις οι επενδυτές. Δηλαδή Βεβαίω εντό τη Ένωση αυτά είναι σαφή. Οι επενδυτέ δεν μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν γιατί υπάρχουν ε, νομοθεσίε. Αλλά ορισμένοι επενδυτέ που επενδύουν σε αδύναμε χώρε, για παράδειγμα, αξιοποιούν την κυρίαρχη θέση του για να χτυπήσουν τα συνδικάτα, για να καταστρέψουν το περιβάλλον. Πώ ε, τοποθετείται η Κομισιόν. Οι επενδυτέ πρέπει να έχουν και υποχρεώσει που ε, να μπορούν να γίνουν απαιτητέ και έναντι του δικαστηρίου αυτό. Και αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων τέλος. Τι αρμοδιότητες και τι καθήκοντα θα έχει έναντι άλλων επιτροπών. Για παράδειγμα, έχουμε τον ε, διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ εξηγήστε μου. Τι συμπληρωματική προστιθέμενη αξία θα σας δώσει αυτή η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαλόντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι απολύτως ε, απαραίτητο να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων και να προβληματιστούμε όλοι για την εξέλιξη της εμπορικής πολιτικής, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην εξέλιξη της δομής των συναλλαγών μας και ώστε αυτή να ανταποκρίνεται επίσης στις προσδοκίες των πολιτών. Έχω ένα προβληματισμό να μοιραστώ μαζί σας και τρεις ερωτήσεις. Η τελευταία συζήτηση για τις εμπορικές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά έδειξαν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν οι συμφωνίες για το εμπόριο να συνάδουν περισσότερο με τις συμφωνίες για το περιβάλλον, να υπάρχουν κανόνες για την δημόσια υγεία, για το δημόσιο αγαθό που πρέπει να καταλαμβάνει μεγαλύτερη θέση. Μπορούμε να επηρεάσουμε την πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, παράδειγμα είναι οι εργασίες της Επιτροπής Σουμπέρ στη Γαλλία Επιτροπή που διατυπώνει κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρουσες ιδέες όπως είναι ένα περιβαλλοντικό βέτο δικαίωμα αρνησή Υπάρχει και ένα κεφάλαιο για την αηφόρο ανάπτυξη που θα πρέπει ίσως να έχει την ίδια νομική ισχύ με τα υπόλοιπα κεφάλαια της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών. Αυτέ είναι οι ιδέε. Τι, είναι ο ρόλος που μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να παίξει για να μετριάσει τι επιπτώσεις τη αρνητική τη παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Ντέβιτ Μάρτι. Δύο ε, παρατηρήσεις κύριε Πρόεδρε, ίσως τρει θα έλεγα. Η πρώτη έχει να κάνει με τη Σιγκαπούρη. Η Αυστραλία και η Νέα Ισλανδία μπορούν να περιμένουν, γιατί μόλι τώρα ξεκίνησε η εντολή διαπραγματεύση, η συζήτηση για αυτή. Αυτό το θέμα είναι πιο επίγοντο συγκεκριμένο. Μιλάμε για το πρώτο γύρο ε, στα τέλη Οκτωβρίου. Πρέπει να πάρουμε απόφαση σύντομα και θα θεωρηθεί προηγούμενο. Ή συζητούμε, ε, ζητούμε από το Συμβούλιο να πάρει απόφαση για τη Σιγκαπούρη με μεμονωμένο τρόπο και να αφήσουμε τα υπόλοιπα για αργότερα. Αν ξανακαθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ, δεν είναι και πολύ πιθανό βέβαια αυτό, θα έχουμε TTIP χωρίς το ΆΗ. Είναι μια ιστορική εντολή. Θα μπορούσαμε να, έχουμε, να βγάλουμε το καμάτι το επενδυτικό, γιατί αυτό ήταν και το πιο ακαθόδες στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Θα ήταν πιο εύκολο δηλαδή αν βγάλουμε αυτό το κεφάλαιο από τις διαπραγματεύσεις. Και τέλος, συμφωνώ με αυτά που είπατε στο τέλος της παρέμβασής σας. Σαφέστατα τα εθνικά κοινοβούλια και στο εμπόριο και γενικότερα έχουν ως ρόλο να κρατούν τους υπουργούς τους υπόλογους. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν αν δεν υπάρχει ροή πληροφοριών και είχαν την πληροφορία αυτή τα κοινοβούλια στη ΣΕΤΑ στο τέλος της διαδικασίας και δεν μπορούσαν να απαιτήσουν λογοδοσία από υπουργούς. Έχετε δίκιο πρέπει τα κοινοβούλια να έχουν το τελευταίο λόγο μόνο αν έχουν διαφάνεια εξ αρχής για να μπορούν οι υπουργοί να είναι υπόλογοι. Άρα με τη δική μας θεσμική δομή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει στα τέλη της διαδικασίας. Πράγματι λέει ο Πρόεδρος, ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο ισχύει αυτό. Μίλησα με περιφερειακού και κυβερνήσει στη Γερμανία και τους κατέστησα σαφές ότι μπορούν να παρέμβουν και να δώσουν εντολή στην κυβέρνησή τους. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν είναι ξεχωριστή αυτή εντολή και πρέπει να δοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, σε διαπραγματεύσεις, πώς θα ταιριάξει με την αρχική εντολή και πώς θα επιταχυνεί το ρυθμό με τον οποίο θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Έχω την εντύπωση ότι πολύ συχνά ε, οι διαπραγματευτές ε, υφίστανται πολύ μεγάλη πίεση για να ε, υποχωρήσουν για θέματα προστασίας επενδύσεων πριν μπορέσουν να διαπραγματευτούν κάτι άλλο. Δηλαδή ο χρόνος πιέζει και δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα αρκετά καλά. πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της επιτάχυσης του ρυθμού των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, μου κάνει ιδιαίτερη ευχαρίστηση αυτή η έκθεση. Δεν θέλω έλεγα ότι είμαι απολύτω ικανοποιημένη, αλλά θεωρώ ότι αποτελεί ένα καλό βήμα προς τα εμπρός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι επιτέλους αναγνωρίζει τις αρνητικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης. Αυτό αποτελεί πρόοδο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει στρέβλωση του εμπορίου, ε, ανηλίκρινες πρακτικές ότι μεγάλες πολυεθνικές μπορούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα χρησιμοποιώντας τη φοροαποφυγή. Πολλά πράγματα δεν πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιτέλους η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι είναι αιτιολογημένος ο θυμός της κοινωνίας και ότι απαιτείται κάποια απάντηση. Αυτό η, η έκκληση της κοινωνίας δεν προέρχεται από το πουθενά και χαίρομαι που το αναγνωρίζει η Επιτροπή. Ωστόσο δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένη διότι πιστεύω ότι η Κομισιόν δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα τι ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει. Εξακολουθεί να θεωρεί ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια θετική έννοια. Τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, ε, κέρδη για τι επιχειρήσει, δουλειέ, ε, καλές για του καταναλωτέ. Θεωρεί ότι είναι εντάξει τα πράγματα, αλλά στο μεταξύ αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ε, ένα πολυμερές δικαστήριο επενδυτικό απλά θα εξυπηρετήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις ε, εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλίματος και των πολιτών. Ε, αυτό δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση. Η Κομισιόν προβλέπει μεγαλύτερη κατανάλωση, αλλά αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη μεταφορά εμπορευμάτων με δυσμενή συνέπειες για το περιβάλλον, λιγότερο ευέλικτη αγορά και πολλά άλλα προβλήματα. θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα υπονομευθεί η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα των προϊόντων. Δεν μπορεί πάντα να έχει κανεί τα φθηνότερα αγαθά και τις φθηνότερε υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρχει ένα κατώτατο όριο κάπου. Και πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη και άλλα θέματα. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η πολιτική αυτή θα, έχει διάφορα ελαττώματα ότι θα οδηγήσει σε προβλήματα για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους και ότι πολλοί ε, δείκτες ε, ποιότητας ε, δεν λαμβάνονται υπόψη όσο θα έπρεπε. Πιστεύω λοιπόν εγώ ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζομένους, περισσότερες διατάξεις για την βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα όσον αφορά την απέτηση συμμόρφωσης με τις κλιματικές απαιτήσει των Παρισίων. Καλό είναι να εστιαζόμαστε στα κέρδη των επιχειρήσεων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την ευημερία των ανθρώπων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι που η Κομισιόν μαθαίνει από τα παλιά της λάθη. Και είμαι περίεργη να δω πώς θα, τι μορφή θα λάβουν όλα αυτά στο μέλλον. Αναφέρεται μια έκθεση που θα βγει το Νοέμβριο για την υλοποίηση των ε, συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών που έχουν συναυθεί μέχρι στιγμής. Θα ήθελα να σας προτείνω το εξής. Ε, βάσει του πνεύματος της ομιλίας του κυρίου Γιούγκερ, ε, όταν αναφέρθηκε στην ε, δημοσίευση των σχεδίων των διαπραγματευτικών εντολών, μπορείτε να μας υποσχεθείτε ότι θα δημοσιευτούν και οι παλιές διαπραγματευτικές εντολές για να γίνει μια σχετική αξιολόγηση. Πιστεύω ότι αυτό θα γινόταν ιδιαίτερα δεκτό και θα ικανοποιούσε πολλού. Μετά τώρα, όσον αφορά τη διαφάνεια, ε, οι συναδέλφοι και ειδικότερο ο David Μάρτιν το είπαν πολύ σωστά. Κάθε εθνικό κοινοβούλιο είναι εκείνο που θα πρέπει να ε, συνομιλήσει με τους υπουργούς του και την κυβέρνησή του. Οι ευρωβουλευτές εδώ και οι πολιτικές ομάδες μάλιστα θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν ε, τα κόμματα στις χώρες τους να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ, όσον αφορά τη συμμετοχή ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εγώ χαίρομαι βέβαια, προέρχομαι από μια χώρα όπου το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά. Τώρα αυτή η ιδέα ότι τα σχέδια εντολής θα, θα πηγαίνουν γρήγορα πριν δημοσιευτούν πολύ νωρί στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένα επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι το εξή. Το Ευρωκοινοβούλιο και ενδεχομένω και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα μπορούσαν να ε, γνωμοδοτήσουν πριν πάει το σχέδιο εντολής στο Συμβούλιο. Μπορείτε να φανταστείτε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να εμπλακεί πιο επίσημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ε, διαπραγματεύσεις ε, αυτές ε, για την εντολή. Φυσικά αυτό θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των όσων επιτρέπουν οι συνθήκες, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιο τρόπος. Τέλος, είδα λίγο την έκθεση υλοποίησή σας για το εμπόριο για όλους. Είναι πολύ σημαντικό μοντέλο ε, που περιλαμβάνει τους στόχους και την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί αναφέρεται ο κανονισμός ε, για τα ε, μέταλλα από περιοχές διενέξεων και τα ορυκτά από περιοχές όπου μένονται σειράξεις. Γιατί διστάζει η Κομισιόν να ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα και σε άλλους τομείς ή σε πιο, πιο ευρεία βάση αυτό το, να, καταστήσει υποχρεωτικό αυτή την επιμέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Είχα κλείσει την λίστα μιλητών, αλλά εντάξει μπορείτε να κάνετε μια σύντομη παρατηρήση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ε, σχημάτισα την εντύπωση κύριε Πρόεδρε Τώρα για το πώς ε, αποφασίζετε ποιοι είναι οι ομιλητές. Ρώτησα στην αρχή ποιος θέλει το λόγο. Δήλωσαν όσοι θέλουν το λόγο και μετά είπα κλείνω κατάλογος ομιλητών. Τώρα με συγχωρείτε αν δεν είδαμε κάποιον ζητάμε συγγνώμη. Οπότε ε, θα δεχθώ να πάρουν το λόγο και οι άλλοι δύο συνάδελφοι. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε αυτή τη μέθοδο. Ποιος θέλει τώρα το λόγο παρακαλώ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Συγγνώμη αν δεν ε, καταλάβατε ότι είχα ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ενημέρωση. Και εγώ θεωρώ ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν ε, περιλαμβάνει ενδιαφέροντα σημεία και ενδιαφέρουσε ε, νέες εξελίξει, αλλά διαφωνώ με ορισμένε σκέψεις. Ε, σε συγχαίρω για τις νέες πρωτοβουλίες όπως το εργαλείο ελέγχου των άμεσων επενδύσεων και τη δημοσίευση των διαπραγματευτικών εντολών, αλλά αντιτίθεμαι για άλλη μια φορά στην ιδέα δημιουργίας ενός πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου. Αλλά θα επιχειρηματολογήσω για να υποστηρίξω τη θέση μου στη σχετική συζήτηση. Το κείμενο υποστηρίζει ότι οι συνθήκες είναι αθώες για τους πολίτες μας. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος διότι έχουμε πολλά παραδείγματα ε, τροποποίησης ή ακύρωσης ευρωπαϊκής ε, νομοθεσίας για να βολευτούν ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και υπάρχουν και παραδείγματα συνθήκων ε, ευρωπαϊκών συμφωνιών που είχαν τελικά αρνητικές επιπτώσεις στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες ε, έχουμε εμπορικές συναλλαγές από ανθρώπους που υποτίθεται ότι προωθούν ισότιμο εμπόριο. Οπότε τη βιώσιμη ανάπτυξη φυσικά χαιρόμαστε που τη συμπεριλαμβάνουμε στις μελλοντικέ συμφωνίες αλλά αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να συνοδεύονται και από για να εξυπηρετήσουν σε κάτι Αλλιώς ε, θα είναι ε, κενά λόγια και δεν θα υπάρχει καμία ε, κύρωση. Όσον αφορά τη συμπερίληψη τη κοινωνία των πολιτών στην εμπορική πολιτική, αναμφίβολα είναι καλό. Θέλω να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ θα γίνει αυτό, πώ θα την πείσουμε. αν εμποδίζονται τα εθνικά κοινοβούλια, πώς θα ακουστεί η κοινωνία των πολιτών. Τώρα όσον αφορά τη δημιουργία του συμβουλευτικού οργάνου, σίγουρα είναι μια καλή ιδέα. Ξέρουμε όμως ότι ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες. Να δούμε λοιπόν αν αυτός ο οργανισμός ε, απλά θα βοηθά στην ε, επικύρωση των αποφάσεων της Κομισιόν ή αν θα συμπεριλαμβάνει και την άψη των ε, πολιτών. Τώρα για τις εμπορικές συμφωνίες με την Αυστραλία, την Νότια Αμερική, ελπίζω η Κομισιόν να ακούσει όλους τους τομείς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη παράγει τρόφιμα και έχει μια γεωργία και αυτοί οι τομείς πρέπει να ε, προστατευτούν ακόμη και αν δεν είναι η πλειοψηφία του όγκου των ε, ε, ανταλλαγών. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ομολογώ ότι δεν είχα, πάρει, δεν είχα ζητήσει το λόγο, αλλά θέλω να σας πω ότι χθε συμμετείχα στην ακρόαση Χόγκαν για τη Γεωργία. Στην ακρόαση του Επιτρόπου Χόγκαν για την Γεωργία, συγγνώμη. Αυτό που με τρόμαξε ήταν η κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις χώρες Μερκοσούρ. Όπως ξέρετε υπάρχουν προβλήματα Απάτη στον τομέα του κρέατος, κυρίως με τη Βραζιλία. Και μετά ε, η πολύ σημαντική ποσότητα πολλών τόνων κρέατος που θα εξαχθεί στην Ευρώπη ε, μέσω της ΕΤΑ ε, έχουν, ε, βρίσκονται σε στασιμότητα οι διαπραγματεύσεις δεν μιλάμε ιδιαίτερα για τη Μερκοσούρ ε, και θέλω να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αλλά και τις προτάσεις τις οποίες θα μεταφέρω στους ε, ανώτερους μου για να τις εξετάσουμε και να τις προωθήσουμε. Ορισμένοι ε, υποβάλλατε τις ίδιες ερωτήσεις. Βεβαίως ε, γίνεται μια συζήτηση και εδώ και αλλού για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τις κυρώσεις. Έχει υποβάλει ένα κείμενο κομισιόν, συνεχίζεται η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα σήμερα να πω τίποτα περισσότερο. Βεβαίως, είναι θέμα συζήτησης και ο Επιτροπός μου και όλη η Γενική Διεύθυνση ξέρει τη σημασία που δίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό, ο διάλογος θα συνεχιστεί. Όμως ε, υπάρχει κάτι ακόμη. Έχει όρια η εμπορική πολιτική. Βεβαίως είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Πιστεύω ότι έχουμε την πιο φιλόδοξη εμπορική πολιτική παγκοσμίω. Αλλά φυσικά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εξωτερική ή άλλες πολιτικές. Υπάρχουν όρια στο τι είναι εφικτό μέσω της εμπορικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να τα φορτώσουμε όλα στην εμπορική πολιτική. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν και όρια. Προοπτική φύλου, ιδιαίτερα για την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Πολύ καλή σύσταση. Σίγουρα στους, ε, στην περιγραφή των καθηκόντων αυτής της νέας ομάδας θα υπάρξει βέβαια ανώτατο όριο ε, του αριθμού των εμπειρονομών, θα είναι 30 ή 40 αλλά νομίζω ότι μια πρώτη αντίδραση στην πρότασή σας είναι πολύ θετική σχέση μεταξύ αυτής της νέας ομάδας και των υπαρχουσών δομών για διάλογο με τους εμπλεκομένους φορείς. Κοιτάξτε, ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών είναι ένας ανοιχτός διάλογος, μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί, δεν αποκλείεται κανείς. Όποιος θέλει να συζητήσει, μπορεί να συζητήσει. Αυτό βέβαια έχει τη δική του αξία, αλλά αυτή η νέα ομάδα θα έχει πιο ολοκληρωμένη δομή για να λάβει η Κομισιόν κάποιες, κάποια βοήθεια που δεν τη λαμβάνει μέσω του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Είχαμε επίσης την συμβουλευτική ομάδα για το TTIP που τώρα δεν λειτουργεί. Άρα δεν θέλουμε να δοθεί εντύπωση ότι έχουμε καταλήψει αυτή τη μέθοδο εργασίας ε, και μας βοηθάει για να δημιουργήσουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους εμπειρογνώμονες να ξέρουν ότι συνεργάζονται σε μόνιμη βάση μαζί μας. Πρέπει λοιπόν να γίνει γνωστή αυτή η πρόσκληση προς εμπειρογνώμονες για να συμμετάσχουν ή να έρθουν οι καλύτεροι. Τώρα, προστασία επενδύσεων. Αναφέρθηκαν διάφορα. Και για αυτό το πολυμερές ε, δικαστήριο για τις επενδύσεις. Αυτό βεβαίως ε, είναι κάτι μακροπρόθεσμο. Δεν θα αρχίσει να λειτουργεί πριν λήξει η παρούσα θητεία τη επιτροπή, αλλά είναι σημαντικό να συνεχίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίζει τον ηγετικό ρόλο στην ε, παγκόσμια συζήτηση για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα με μεγάλες δυσκολίες. Και γι' αυτό τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι για συμφωνίες με χώρες όπως ε, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζεται καν τέτοιο δικαστήριο γιατί αυτές είναι χώρες όπου λειτουργεί το, το κράτος δικαίου. Οποιοδήποτε έχει πρόβλημα μπορεί να απευθυνθεί στα δικαστήρια. Αλλά το αντιπιχείρημα είναι τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ χωρών. Για παράδειγμα στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα χρειαζόμαστε ένα δικαστήριο προστασία των επενδύσεων. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιο στην συμφωνία με την Αυστραλία, θα έχουμε πρόβλημα. Κάποιο τέτοιο δικαστήριο. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω πολύ περισσότερα. Πώς θα πάμε τώρα στη διαπραγματεύση με τη Σιγκαπούρη. Είναι διαδικασία ε, αναδιάρθρωσης της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με τη Σιγκαπούρη. Είναι μεικτή η συμφωνία όπως τη λέμε εμείς γιατί υπάρχει ένα τμήμα για την προστασία των επενδύσεων. Τώρα θέλουμε να ε, διαχωριστεί από την υπόλοιπη εμπορική συμφωνία και να υποβληθεί χωριστά. Βλέπουμε ότι η Σιγκαπούρη ε, το αντιμετωπίζει θετικά. Βέβαια πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Προχωράνε λοιπόν ε, και ελπίζουμε να σας υποβάλουμε ε, στις αρχές του επόμενου χρόνου και σε εσά και στο Συμβούλιο την συμφωνία για την επίσημη ε, έγκριση. Αλλά αυτή είναι η προτεραιότητά μας μαζί με το Βιετνάμ, όπου η κατάσταση είναι παρόμοια. Οι διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ όμως ε, δεν προχωράνε τόσο γρήγορα όσο με τη Σιγκαπούρη. θα υπάρξουν δύο στιγμές αληθείας πολύ σύντομα. Η πρώτη θα είναι όταν ε, το Συμβούλιο και εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε τις δύο συμφωνίες με την Σιγκαπούρη ή όταν το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις για την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Τότε θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το διαχωρισμό της αντιμετώπισης ε, για την προστασία των επενδύσεων. Έχουμε κάνει πολλέ συζητήσει ε, πρόσφατα στο Τάλιν, πριν από δύο εβδομάδες. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να υιοθετήσουν τελική στάση χωρίς να υπάρχει και μια συγκεκριμένη διατυπωμένη πρόταση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει λοιπόν τις συγκεκριμένες προτάσεις και μετά θα δούμε πώς θα αντιδράσουν τα κράτη-μέλη. και αν ε, ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το TTIP ε, ή για κάποια άλλη παρόμοια συμφωνία, βεβαίως θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας, για την προσέγγισή μας, για τις σχέσεις και την εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι ο μόνος τρόπος ε, για να επιτύχουμε. Βεβαίως. Και εμείς ως Γενική Διεύθυνση Εμπορίου πολύ συχνά έχουμε κάθε κατανόηση για τις επικρίσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών ή των κοινοβουλίων. Δεν είναι ότι είμαστε κλεισμένοι σε χρυσελεφάντινο πύργο, αλλά δεν είναι δυνατόν μια γενική διεύθυνση 600 ε, συνεργατών να τα επιτύχει όλα αυτά εργαζόμενοι από τις Βρυξέλλες. Πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς, τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση κυρία Μακλάρκιν. Αναφερθήκατε σε μία άλλη σημαντική διάσταση της προστασίας των επενδύσεων. Βεβαίως, γίνονται χωριστά διαπραγματεύσεις και υπάρχουν ενδεχομένως και δύο εντολές για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Μάλλον έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Όταν θα έχουμε μια σαφή εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί η προστασία των επενδύσεων, εάν θα παραμείνει τμήμα κάθε συμφωνίας ελευθερού εμπορίου, τότε θα είναι πιο απλή κατάσταση γιατί οι διαπραγματεύσεις ε, θα διεξάγονται παράλληλα και για τις δύο αυτές ε, συμφωνίες. Εάν τελικά θα καταλήγουμε σε δύο διαφορετικές συμφωνίες, αυτό δεν επηρεάζει την διαπραγματευτική μας τακτική, όπως σωστά είπατε. Θα πρέπει ορισμένες απρόθυμες ε, τρίτες χώρες να λάβουν κάποιες παραχωρήσεις ε, στη Συμφωνία Ελευθερωμπορίου για να συμφωνήσουν μαζί μας για την, ε, το μηχανισμό ε, διαφορών. Αυτό είναι δικό μας εσωτερικό θέμα. Δεν, ε, δεν έχει επιπτώσει στην χώρα με την οποία διαπραγματευόμεθα. Αλλά παρόλα αυτά αυτό που είπατε ισχύει. Θα μιλήσω λοιπόν τώρα τη γλώσσα μου. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Σα, σας ευχαριστώ πολύ και να πω το εξής που θα ήθελα να σημειωθεί. Η, η Κομισιόν δεν νομίζω ότι προτείνει εξίσωση προς τα κάτω. Όχι. Στόχος μας είναι να υπάρξει μία πρόοδος προς τα άνω, ούτως ώστε να ε, εξαχθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρότυπα. Σίγουρα δεν επιδιώκουμε αυτό που είπατε. Δεν ανταποκρίνεται στο πώς ε, αντιμετωπίζω το θέμα και πώς αντιμετωπίζει η υπηρεσία μας ε, το θέμα. Νομίζω ότι το υπόδειγμα της Φιλανδίας και των σκανδιναβικών χωρών είναι θετικό, καλό θα ήταν να επεκταθεί και σε άλλα κράτη-μέλη που δεν είναι τόσο δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στην εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μπορεί, μπορεί το Κοινοβούλιο να εμπλακεί στην διατύπωση της διαπραγματευτικής εντολής. Η Επιτροπή και οι υπάλληλοι μας πάντα σας ακούμε. Είμαστε εδώ και είμαστε υπόλογοι σε εσά. Φυσικά κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ε, εντολής λαμβάνουμε υπόψη αυτά που μας λέτε αλλά ε, θεσμικά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επίσημη εμπλοκή της Επιτροπής σας πριν διατυπώσουμε το σχέδιο διαγωνιστικής εντολής. Για το Μερκοσούρ, κύριε Φεράν, χθε συμμετείχα σε μια συνεδρίαση άνω των δύο ωρών στην Επιτροπή Γεωργίας για το Μερκοσούρ για το θέμα του βοήου και της εθανόλης. Παρουσίασα όλα τα επιχειρήματα για να υποστηρίξω αυτή την ε, προσφορά, αλλά δεν νομίζω ότι έπεισα πολλούς και ιδιότερα βεβαίως όχι την πολιτική σας ομάδα. Ωστόσο, δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε συζήτηση για το Μερκοσούρ. Ε, με χαρά να έρθω ή εγώ ή κάποιος άλλος κάποια άλλη στιγμή να το συζητήσουμε. Αλλά δύο σημεία είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να είναι σαφή για όλους. Αν δεν υπάρξει ουσιώδης ε, προσφορά για το βόιο και την εθανόλη, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Αυτό είναι σαφές. Όσοι λένε ότι πρέπει να εξαιρεθεί το βόιο και η εθανόλη, στην ουσία λένε δεν θέλουμε Μερκοσούρ. Εντάξει, είναι μια άποψη, αλλά δεν είναι η δική μα. Ούτε ως Κομισιόν, ούτε ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, στην παρουσίαση τη προσφορά που θα κάνουμε την προσφορά που καθυστέρησε ένα χρόνο. Επειδή ήταν πολύ λεπτό το θέμα αυτό, καθυστερήσαμε. Θέλαμε να γίνουν σημαντικές εκλογές πρώτα στην Ευρώπη. Ο τρόπος παρουσίας της προσφοράς μας λαμβάνει υπόψη τις διάφορες ευαισθησίες. Ιδιαίτερα έχοντας ε, την προσφορά σε δύο τμήματα. Το 1 τρίτο της ε, βιοεθανόλης το 1 τρίτο τη Αθανόλη που προτείνουμε να δεχτούμε είναι βιοεθανόλη και τα άλλα 2 τρίτα είναι μόνο για ε, βιομηχανικέ χρήσει. Και για την. Ε, και για το βόλιο έχει δύο τμήματα η προσφορά μα, 35.000 κατεψυγμένα, 35.000 τόνοι πάντα, φρέσκο. Νομίζω ότι έτσι λαμβάνουμε υπόψη όλε τι ευαισθησίε που υπάρχουν στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Θα παραμείνουμε σε επαφή. is on our... Και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τα θετικά και τα αρνητικά της παγκοσμιοποίησης. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ πολύ. Good. Die nächsten beiden Punkte. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι επίση ένα σημαντικό στοιχείο τη εμπορικής πολιτικής. Το μέλλον του ΠΟΕ, το σημείο 6. Μία αντιπροσωπεία μας πήγε στη Γενέβη για ένα δημόσιο φόρουμ στις 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Είναι μια καλή παράδοση αυτή, αυτό το δημόσιο φόρουμ όπου γίνεται δημοσίω γνωστή η εργασία του ΠΟΕ και συζητείται με την κοινωνία των πολιτών. Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με, ε, το IPU, διοργανώσαμε μία εκδήλωση για το πώς μπορεί να είναι δίκαιο το εμπόριο, πώς θα καταστήσουμε δίκαιο το εμπόριο. Τοποθετήσαμε εκεί την ε, κοινοβουλευτική προοπτική, είχαμε πολύ καλή συμμετοχή, συνολικά συμμετείχαν 2.000 ε, σε αυτό το δημόσιο φόρουμ σε 150 διαφορετικές εκδηλώσεις. Ήταν μια, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για να γίνει γνωστή η λειτουργία του ΠΟΕ που μέχρι στιγμής δεν ήταν καθόλου γνωστή. Ήταν παρούσα η κυρία Λαγκάρντ, η Υπουργός της Αργεντινής ε, κυρία Λακόρα και ο κύριος Κρούκμαν. Ο Κρούκμαν που είναι γνωστός από τα μέσα. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Όπως είναι σύνηθες, συζητήσαμε και με συναδέλφους από άλλα κοινοβούλια για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον του ΠΟΕ στην ε, μόνιμη επιτροπή της ε, κοινοβουλευτικής διάσκεψης. Στόχος μας ε, είναι βεβαίως τελικά να ελέγχεται και κοινοβουλευτικά εργασία του ΠΟΕ και να υπόκειται στις, στους αναγκαίους περιορισμούς. Αυτός είναι ο στόχος της κοινοβουλευτικής διάσκεψης. Και στόχος μας ήταν πρώτα απ' όλα η προετοιμασία της υπουργικής ε, συνάντησης στο Μπουένος Άιρες. Οι οργανωτικές ε, προετοιμασίες πάνε καλά. Οι ουσιώδεις προετοιμασίες, δηλαδή για το τι θα συζητηθεί, επηρεάζονται από την ε, αβεβαιότητα για το τι θα κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον πρέσβη της Ένωσης και ορισμένους άλλους ε, σημαντικούς πρέσβης που έχουν μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση για το μέλλον του ΠΟΕ και θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα προς αυτή την κατεύθυνση. συμμετείχαν η Ίνμα και η ΕΜΑ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα. Έμα, όχι. Καλά. Ωραία. Θα σας διανεμηθεί και μία γραπτή έκθεση. Και να μπορέσετε να διαβάσετε τι έγινε. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 7, το οποίο συνδέεται. Όπως είναι γνωστό, ε, θα λάβει χώρα 10 με 13 Δεκεμβρίου η 11η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Πένο. Άιρες. Ως Κοινοβούλιο θα εκπροσωπηθούμε μέσω 15 μελούς αντιπροσωπείας ως μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας της Ένωσης. Σημαντικό αυτό. Εμείς ως Κοινοβούλιο βεβαίως έχουμε απέτηση να παρακολουθούμε και να συνοδεύουμε και να ελέγχουμε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ε, που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπάρχει μια σαφής εντολή. Ως ε, συμπρόεδροι της ε, Διοικητικής Επιτροπής, ο κύριος ε, Ρούμπιχ και η ταπεινώτε μου, σας υποβάλαμε ένα σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο πριν τη διάσκεψη θα εγκριθεί και από την Ολομέλεια. Ούτως ώστε να υπάρχει σαφής κατεύθυνση για το ποια θεωρούμε εμείς ότι είναι τα κεντρικά σημεία που θέλουμε να συμπεριληφθούν στις συζητήσεις. Είμαι πεπισμένο ότι δεν θα είναι απλές οι εργασίες αυτή της διάσκεψης. Και σε άλλα σημεία τη σημερινής διάταξη αναφερθήκαμε στην ε, συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ξέρετε στο Μαρακές υπήρξε μια προπαρασκευαστική διάσκεψη, μια άτυπη συνάντηση ορισμένων υπουργών και, επιτρόπου, και της Επιτρόπου. Ο κύριος Λάιτχάιζερ, ο Αμερικανός ε, εντεταλμένος για το εμπόριο, την τελευταία στιγμή ακύρωσε τη συμμετοχή του. Αυτό καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούν ενεργά οι Ηνωμένε Πολιτείε σε αυτή τη συγκυρία με τον ΠΟΕ. Γι' αυτό είναι σημαντικό εμείς μαζί με τους άλλους εταίρους να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε να διατηρήσουμε εν ζωή θα έλεγα το παγκόσμιο εμπόριο και να επιτύχουμε και κάποιες περαιτέρω πρόοδους. Βέβαια δεν θα επιτύχουμε τίποτα το τρομερό. Πρέπει ωστόσο να κάνουμε έντονο διάλογο με τους εταίρους μας ε, επί του εφικτού. Από ό,τι φαίνεται και οι αναπτυσσόμενες χώρες ανησυχούν ιδιαίτερα για την έλλειψη προόδου για την εφαρμογή του θεματολογίου της ΔΟΑ. Οπότε αυτή η διάσκεψη του ΠΟΕ ίσως και να μην επιτύχει. Οπότε, το καθήκον ημών των κοινοβουλευτικών από όλα τα κοινοβούλια είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να μην καταρρεύσει το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Πριν από τη διάσκεψη, στις 19 Δεκεμβρίου, θα λάβει η χώρα μια κοινοβουλευτική συνάντηση. Και αυτό πρέπει να είναι το μήνυμά μας. Θέλουμε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα που να βασίζεται σε αξίες. που να βασίζεται σε αρχές δικαίου και όχι στο δίκαιο του χειροτέρου. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου. Θέλει κανείς το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε να μας μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση Εμπόριου. Ο κύριος Πιτοάρη Ντετσκόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω δύο λόγια για την ε, κατάσταση των προετοιμασιών και της 11 η Υπουργικής Συνόδου και το τι συνέβη στο Μαρακές τις τελευταίες ημέρες. Δευτέρα και Τρίτη πολλές υπουργικές συναντήσεις έλαβαν χώρα, συμμετείχαν περίπου 40 υπουργοί και συζήτησαν σε βάθος ε, τις προετοιμασίες της 11ης Υπουργικής Συνόδου. Σε αυτή την Υπουργική Διάσκεψη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσώπησε η Επίτροπος Μάιλστρομ, η οποία επανέλαβε την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη η Υπουργική Διασύνοδος να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, να γνωρίζουμε τη δουλειά που έχει γίνει σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις στην αλία και τα αποθέματα για λόγους ε, επισητιστικής βοήθειας τροφίμων, ε, υπαρκούς ε, αποθεμάτων τροφίμων. Πολλά ζητήματα προετοιμάζονται Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με αυτά τα δύο ζητήματα, πρέπει να ασχοληθούμε και με περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες για να φτιάξουμε ένα πακέτο στον Buenos το οποίο να είναι ισορροπημένο συγκεκριμένες αποφάσεις, συγκεκριμένα αποτελέσματα ισορροπία μεταξύ αυτών και ισορροπία μεταξύ αυτών και της μελλοντικής δουλειάς στο πλαίσιο του ΠΟΕ μετά την Υπουργική Σύνοδο στον Πόνος Άιρες. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση κάναμε διάφορες προτάσεις για τη δουλειά για τους επόμενους μήνες, εγχώρια στήριξη στη Γεωργία για παράδειγμα. Αυτό είναι σημαντικό για πολλά μέλη και συνδέεται άρεκτα με τα public stock holdings για λόγους επάρκειας τροφίμων. Κάναμε δουλειά για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για τον εγχώριο κανονισμό, για τις υπηρεσίες, για τη διαφάνεια στο ε, ANTB, για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις ενισχύσεις στη βιομηχανία. Παρόλο που η συζήτηση στο Μαρακές ήταν δύσκολη και περίπλοκη, πρέπει να υπογραμμίσω ότι οι δεσμεύσει είναι σημαντικέ. σημαντικές. Πολλά κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα αιτήματα για διάφορα θέματα, όπως τα μη δεσμολογικά εμπόδια. Βέβαια υπάρχουν αποκλήσει μεταξύ των μελών για τα θέματα στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει πραγματική πρόοδος. Όλα αυτά τα συνόψε σωστά ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕΣ χθες το απόγευμα, ο οποίος είπε ότι υπάρχει φιλοδοξία αλλά δεν υπάρχει ακόμα ρεαλισμός και χρειάζονται και τα δύο. Ο Υπουργό Εμπορίου του Μαρόκο προείδρευε και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση αναφερόμενος στους εξής τομείς συνεργασίας που θεωρεί ότι έχουν προοπτικές. Πρώτον, γεωργία. Δεύτερον, ενισχύσει στην αλία. Τρίτον, χώροι κανονισμοί για τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών. Και τέλος, συνέχιση της συζήτησης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, διότι αυτό είναι σημαντικό για πολλά μέλη. Τέλος, ο Υπουργός Μαλκόραν πρόεδρος της Υπουργικής Διάσκεψης στο Buenos ολοκλήρωσε συνόψισε λέγοντας ότι το πακέτο που θα πρέπει να τύχει αντικείμενο συμφωνίας MC11 πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα αποτελέσματα αλλά και στοιχεία που να αποτελούν φυγή προς τα εμπρός ε, και ως προς τις ενισχύσεις και ως προς τη διαδικασία. Προετοιμάζοντας λοιπόν την Υπουργική Σύνοδο, αυτά έχω κυρίως να πω και θα σας στείλουμε ενήμερους και περιμένουμε να έχουμε και καλό συντονισμό επιτόπου στον Πανοσάρις για να υπάρχει επαρκή ροή πληροφοριών και να γνωρίζουν όλοι από πρώτο χέρι τις εξελίξεις στις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Για να είμαι ειλικρινής, η παρουσίασή σας δεν συνάδει με τα στοιχεία που έχω εγώ ε, λάβει από το Μαρακές. Άκουσα ότι είναι πολλές οι συγκρούσεις και δεν μου μετέφεραν καθόλου τον αισιόδοξο τόνο που εσείς μεταφέρατε από πλευράς ε, Προεδρίας. ή τουλάχιστον ο αισιόδοξο τόνο τη προεδρία ίσω είναι μη ρεαλιστικό σε σχέση με τα τεκτενόμενα και σε σχέση και με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τα θέματα που τέθηκαν ή δεν τέθηκαν. Μπορείτε αυτά να τα σχολιάσετε παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Όπως είπα στην παρουσίασή μου προλίγου, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στις συζητήσεις στο Μαρακές. Όμως, Κατά κύριο λόγο, αυτό που έχει μπει στο τραπέζι και αυτό που τα μέλη ε, βλέπουν ότι μπορούν να συγκλίνουν πάνω σε αυτό είναι πιο ότι δηλαδή πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά τις επόμενες εβδομάδες για να έχουμε συγκεκριμένο αποτέλεσμα για τις ενισχύσεις για την αλία και public stock holdings και συμμετοχές για λόγους food security για να υπάρχει συνέχεια σε αυτά που συμφωνήθηκαν στο Ναϊρόμπι. Η Προεδρία λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο περαιτέρω δουλειά στη Γεωργία και στην Αλία και αυτό αποτέλεσε μέρος των συμπερασμάτων του Προέδρου. Μία δίκαιη αξιολόγηση ε, είναι αυτή που έκανε ο Πρόεδρος, ότι δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να γίνει περαιτέρω δουλειά για το κανονισμό για τις υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ε, δύσκολο και ακαθόδες για πολλά μέλη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κείμενο πάνω στο τραπέζι που πάνω από 40 μέλη του ΠΟΕ στηρίζουν είναι περισσότερο θέμα τακτικής, δεν υπάρχει θέμα επί της ουσίας. Και θα μπορούσαν να γίνουν κάποια ε, βήματα. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο τώρα το ζήτημα είναι βασικά πολιτικό. Θα είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στην Υπουργική Σύνοδο στοχεύουμε στο να έχουμε κάτι συγκεκριμένο, συγκεκριμένη δέσμευση, να συνεχιστεί η δουλειά μετά τον Buenos Aires, τουλάχιστον αυτό δηλαδή να πάρουμε. Αυτός ο τομέας ε, είναι αναπόσπαστο μέρος των εργασιών αυτού του οργανισμού και αποτελεί μέρος της μελλοντική ισορροπίας ε, θεμάτων που εξετάζονται. Τώρα, ως προς το ερώτημά σας για τις Ηνωμένε Πολιτείες θα τόνιζα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε στη δήλωσή τους στο Μαρακές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να υπάρχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα στην Υπουργική Διάσκεψη, ωστόσο τόνισαν ότι σε ό,τι της αφορά δεν βλέπουν να υπάρχει μεγάλη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών για άλλα ζητήματα και κυρίως ως προς το ενδεχόμενο να έχουμε φιλόδοξα αποτελέσματα για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Φυσικά, αυτό δημιουργεί πρόβλημα, πράγματι, και είναι κάτι που θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης. Από τη δική μου προοπτική, οπτική γωνία, εμείς πρέπει να μεριμνήσουμε να συνεχιστεί η συζήτηση και να ασκούμε πίεση στους εκάστοτε τομείς ξεχωριστά έτσι ώστε να υπάρχει στους εκάστοτε τομείς όσο δυνατόν περισσότερη τεχνική προόδος. Και άρα θα πάμε στο Buenos Aires με βάση, για, με βάση υπαρκτή για να υπάρχει πραγματική απόφαση ισορροπημένη με συγκεκριμένο αποτέλεσμα και έκβαση και να μην εσωτερικεύσουμε τις αρνητικές ε, ε, απόψεις ε, που εκφράζονται και επιδιώκονται από ορισμένου. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Όπως πολύ σωστά λέγεται, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Παρ' όλα αυτά, θα υποβάλουμε το ψήφισμά μας, τροπολογίες μέχρι τις 17 Οκτωβρίου. Και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 9 Νοέμβριο. Ε, συγγνώμη, ναι, ναι, νοέμβριο. σωστά, ναι. Ε, τι θέλετε να πείτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήρθα καθυστερημένα. Ήμουν σε μια άλλη επιτροπή. Έχετε ήδη συζητήσει τον Buenos Αν έχετε κάποιο σχόλιο, λέει ο Πρόεδρος, σε δύο λεπτά, δύο λεπτά σας δίνουμε. Ο κύριος Στάκουλα. Θα προσπαθήσω λοιπόν από κάτι. Αλλά όπως ξέρετε... Λείπει η ατζέντα και τα μέλη του που αποφάσισαν ε, πρέπει να αποφασίσουν τι θα γίνει για την MC11 για να προλιάνουμε το έδαφος. Δυστυχώς η ατζέντα δεν είναι έτοιμη και τα μέρη δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει για τα διάφορα γεωργικά ζητήματα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτά είναι κάποια πιθανά θέματα όπου μπορούμε να περιμένουμε κάποια αποτελέσματα. Κάποια μέλη δεν φαίνεται να θέλουν να δεσμευτούν ιδιαίτερα για τις επερχόμενες συζητήσεις. Ελπίζω να έχουμε μια ανοιχτή και επικοδομητική συζήτηση με τους άλλους συναδέλφους μας στην 11η Υπουργική Συνάντηση στον Πονοσάιρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις συζητήσεις αυτές, να παίξει κεντρικό ρόλο στον Πονοσάιρες. Θα πρέπει να εχει ενεργο ρολο στη συζητηση αυτες να παιξει κεντρικο ρολο στον πονοσαιρες θα πρεπει να διατηρησουμε το διάλογο και με άλλα μέλη όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία που ενδεχομένως να μην έχουν ε, φιλόδοξους στόχους για την 11η Υπουργική Συνάντηση όπως εμείς. Φυσικά είμαστε οι πιο σημαντικοί στη συζήτηση αυτή. Ε, έχει αναβληθεί ο διορισμός του πρέσβη στη Γενέβη. Ε, η Γεωργία εξακολουθεί να παραμένει το πλέον ευαίσθητο θέμα των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει η Γεωργία στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ε, μου απομένουν 15 δευτερόλεπτα μέσα στα οποία θέλω να πω ότι Ε, ε δεν, αυτά που δεν υπόθηκαν στο Νερόμπι ε, ευελπιστώ να συζητηθούν στο Buenos Aires. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζουμπί, καταρχάς ε, ευχαριστώ και συγγνώμη γιατί ψηφίζαμε στην Ήτρε και γι' αυτό δεν ήμουν εδώ. Ε, έτσι έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς δεν μπορώ να κοπώ στα δύο. Η συνάντηση του ΠΟΕ που επίκειται στο Μπουένος Άιρες είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Τονίζω ότι πρώτα θα γίνει η κοινοβουλευτική συνάντηση. Είναι μια ιδέα που προέκυψε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να συζητήσουμε από κοινοβουλευτική άποψη και τη διοργανώνουμε μαζί με τη Διεθνή Κοινοβουλευτική Ένωση της Γενέβης. Διότι ε, βεβαίως αυτά που συζητούνται στον ΠΟΕ πολλές φορές συζητούνται μετά και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που έχουν λιγότερες δυνατότητες να ενημερωθούν. Θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι στο Buenos Aires θα υπάρξει πρόοδος στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce, κάτι που είναι μεγάλη πρόκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι και στον τομέα αυτό δίδονται πολλές δυνατότητες απασχόλησης γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα επιτύχουμε και για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να τους προωθήσουμε και τους 17 αυτούς στόχους ε, παράλληλα, αλλά θα πρέπει το Κοινοβούλιο να δει ποια θέματα είναι πιο σημαντικά για την Ευρώπη για να τα θέσουμε στην ημερήσια διάταξη. Οπότε, πιστεύω ότι και στα πλαίσια του ΠΟΕ, ως κοινοβουλευτικοί, να θέσουμε τις προτεραιότητές μας που εντάσσονται στη δραστηριότητα του ΠΟΕ και που θα μας επιτρέψουν, πιστεύω, να επιτύχουμε πρόοδο. Γι' αυτό ε, αναμένω ε, με ιδιαίτερη αγωνία να δω πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Όπως είπα και προηγουμένως, τροπολογίες μέχρι τις 17 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου και κατόπιν θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε το ψήφισμα στην Ολομέλεια πριν την ε, συνάντηση του ΠΟΕ θα συζητήσουμε στις 25 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο τα αποτελέσματα της συνάντησης στο Μαρακές. Και τώρα θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή, δύο λεπτά, γιατί το επόμενο θέμα είναι και κλεισμένο των θυρών. Μόνο οι συνήθεις ύποπτη δηλαδή επιτρέπεται να συμμετάσχουν.